Παρουσίαση εκ μέρους του Συμβουλίου της θέσης του σχετικά με το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού Οικονομικό έτος 2016 να δώσω το λόγο στον κύριο Γκραμενά εξ του Συμβουλίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο προπολογισμού της Ένωσης για το 2016 το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου. Ο βασικός στόχος είναι να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη, τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αφενός, καθώς επίσης και να δώσουμε κίνητρα για τη χρηματοδότηση των μεταναστευτικών πολιτικών της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφετέρου. Ο προϋπολογισμός λοιπόν αντικατοπτρίζει την αλληλεγγύη εκ των έσω και την αλληλεγγύη ε, έξωθεν. Θα σας κάνω μία παρουσίαση σε τρία τμήματα. Ε, το πρώτο τμήμα ε, είναι αφιερωμένο στην επικαιρότητα. Ένα δεύτερο τμήμα αφορά τις επτά βασικές αρχές που διέπουν την απόφαση του Συμβουλίου και υπάρχει ένα τρίτο τμήμα ε, που έχει τις ε, λεπτομέρειες. Ε, βλέποντας την τραγική επικαιρότητα με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν από τον πόλεμο και εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην Ευρώπη ε, θεωρώ ότι πρέπει να επισημαίνω την υποστήριξη που ε, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση αυτή τη στιγμή, ε, που έρχεται να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών της Ένωσης. Η κρίση των προσφύγων που ζητούν άσυλο αποτελεί τμήμα της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλεγγύης μας. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Τα δύο βασικά ταμεία ε, που έχουν την επιμερισμένη διαχείριση είναι το Ευρωπαϊκό ε, Κοινωνικό Ταμείο και το ΜΥΦ, τα οποία έχουν 3,1 δις ευρώ και 3,7 δις ευρώ ε, για το 2014-2020 αντίστοιχα. Το 2015 εγκρίθηκαν πάνω από 45 εθνικά προγράμματα ε, αξίας ε, ε, κάτι παραπάνω από ένα δί σε δεσμεύσεις. Έχουν ήδη δοθεί 210 εκατομμύρια σε προχρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την κατεπίγουσα βοήθεια έχουμε αποδεσμεύσει κάτι παραπάνω από 60 εκατομμύρια. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Μάιο του 2015 ενέκριναν την, ε, το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση με τους τέσσερις πυλώνες για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και εγκρίναμε επίσης και τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 5 για το σκοπό αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους βασικούς ε, ε, χορηγούς στην γείτονα περιοχή της Συρίας. 855 ε, εκατομμύρια ανθρωπιστικές βοήθειες έχουν δοθεί στους πρόσφυγες τη Συρία, τη Ιορδανία και τη Τουρκία για το 2016 και η επανεγκατάσταση των προσφύγων είναι στα 150 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα και την Ιταλία για τη βοήθεια στους πρόσφυγες και έγιναν πλήρως αποδεκτά τα ποσά αυτά από το Συμβούλιο. Τα θέματα αυτά ε, σίγουρα θα συζητηθούν αύριο από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ζαν Κλοντ Juncker, ε, στην παρουσίαση της ε, κατάστασης της Ένωσης, όπου θα σας παρουσιάσει μεταξύ άλλων και μια νέα δέσμη μέτρων για τον τομέα αυτό. Το δεύτερο τμήμα αφορά τις επτά βασικές αρχές που διέπουν τις εργασίες του Συμβουλίου. Καταρχάς, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε και να ρυθμίσουμε το θέμα των καθυστερήσεων πληρωμών που θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί μέχρι το τέλος του 2016 και η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει και κατάλληλες πιστώσεις για να ξεκινήσουν οι πληρωμές για το 2015 και το 2016 που καθυστερούν. Δεύτερη αρχή, το Συμβούλιο έχει διατηρήσει το σύνολο όλων των χρηματοδοτήσεων που προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων το 2016 που είναι απόλυτη προτεραιότητά μας. Τρίτον, η μεταναστευτική πολιτική έχει αντίστοιχη χρηματοδότηση. Κάποια προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελλάδος και της Ιταλίας για τη μετεγκατάσταση των 40.000 προσφύγων ε, που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Και επίσης ε, 515 εκατομμύρια ευρώ ε, προοδευτικά ε, για το 2016 σε σχέση με το 2015 και επίσης η ανθρωπιστική βοήθεια. Αυξάνεται κατά 16% το 2016 βοήθεια σε σχέση με το 2015, ποσό το οποίο αναλογεί σε πάνω από ένα δις ευρώ. Οι μειώσεις πιστώσεων που έχουν γίνει εμπνέονται από τις εξής παραμέτρους ε, πρόοδο κάποιων προγραμμάτων, ε, κάποιες εκτελέσεις οι οποίες έχουν εκπνεύσει και έχουν καθυστερήσει και καθώς επίσης τη δυνατότητα απορρόφησης η οποία θα πρέπει να είναι ρεαλιστική για τα διάφορα προγράμματα. Μια έκτη αρχή οι τίτλοι προπολογισμού που έχουν προσαρμοστεί από το Συμβούλιο είναι οι μόνοι τίτλοι για τους οποίους είχε ε, προτείνει πολύ μεγάλη διαφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επρόκειται για ποσά τα οποία ήταν πολύ αυξημένα και σε αυτά έγιναν κάποιες διορθώσεις προς τα κάτω. Αλλά αν δείτε την ε, απόλυτη αύξηση των ε, πιστώσεων στον τομέα αυτό θα δείτε ότι υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις. Έβδομη και τελευταία αρχή επειδή υπάρχει πολιτική αστάθεια και ορισμένες φορές ε, κάποια δραματικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει κατάλληλο περιθώριο ευελιξίας για να μπορέσει να δράσει σε περίπτωση που υπάρχουν ε, αύξηση των εντάσεων και των ε, συγκρούσεων. Και τώρα, πολύ σύντομα, να περάσω λίγο στις λεπτομέρειες της θέσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου ομόφωνα. Προτείνουμε δεσμεύσεις ε, ε, υποχρεώσεων 153,3 δις ευρώ και ε, πληρωμών 142,1 δις. Έχουμε 0,6% αύξηση για τις υποχρεώσεις και μείωση 0,54% γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει μείον 0,5% άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά. Η θέση μας μας επιτρέπει να μειώσουμε τη διαφορά μεταξύ των δεσμεύσεων των υποχρεώσεων και των πληρωμών, τα ε, λεγόμενα υπόλοιπα προς καθάριση, τα ραλ και επομένω μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο τις πληρωμές μας. Όσον αφορά τώρα τις υποχρεώσεις μας ανατίτλο, στον τίτλο της ανταγωνιστικότητας για την, και την, για την ανάπτυξη και την απασχόληση που είναι από τις βασικές προτεραιότητες για τις επενδύσεις και την απασχόληση αυξάνεται κατά 8,6% ε, στις πληρωμές και 7% στις υποχρεώσεις. Για να υλοποιήσουμε το ε, Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων, που είναι απόλυτη προτεραιότητα, έχουν γίνει κάποιες ε, αλλαγές στα εξή θέματα, στο Νορίζοντα 2020 και στο Connecting Europe Facility. Και υπήρξε κάποια μίεση επίσης στα μεγάλα προγράμματα υποδομών, τον Γαλιλαίο, το Ίτερ και το Κοπέρνικους δηλαδή και τις ε, συμπράξεις, ε, στις κοινές συμπράξεις. Παρά τις ε, μειώσεις, το ποσό για τον ορίζοντα 2020 από το 9,3% πηγαίνει στα 140 εκατομμύρια και έχουμε 9,9% σημαντική αύξηση. Επίσης, έχουμε κάποιες μειώσεις στο μηχανισμό για την διασύνδεση για την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, έχουμε αύξηση κατά 5,3% στα 760 εκατομμύρια ευρώ και 203 εκατομμύρια ευρώ για τις πληρωμές, ε, που είναι 14% αύξηση, ε, που είναι σημαντικότερο ποσό. Τα προγράμματα κόσμε και Erasmus τα οποία είναι πολύ σημαντικά, δεν επηρεάζονται από μειώσεις και να σας πω ότι το πρόγραμμα Erasmus Plus έχει 1,8 ε, δις ευρώ για το 2016 που σημαίνει ότι έχουμε αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση με το 2015 στα θέματα συνοχής και οικονομικής και εδαφικής συνοχής ε, μια πολύ μικρή μείωση κατά 0,45% στη βιώσιμη ανάπτυξη φυσικούς πόρους, ε, μικρή μείωση κατά 0,45% των πληρωμών και 0,32% για τις υποχρεώσεις σε σχέση με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον τίτλο 3, ασφάλεια και ηθαγένεια, ε, στον οποίο στάθηκα ήδη στο πρώτο τμήμα της παρουσίασής μου, έχουμε πολύ ισχυρή αύξηση σε σχέση με το 2015, κατά 8,7% στις ε, υποχρεώσεις και πάνω από 15% για τις πληρωμές. Ουσιαστικά εδώ έχουμε τις δράσεις στον τομέα της μετανάστευσης που αποτελούν πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο επίσης δέχτηκε την κινητοποίηση του Ταμείου Ευελιξίας. Στον τίτλο 4, το Συμβούλιο σε μεγάλο βαθμό δέχεται τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έχουμε αύξηση κατά 22,4% για τις πληρωμές, ε, περίπου 9 δις ευρώ. Και εδώ θα ήθελα να σας ε, τονίσω ότι το Συμβούλιο ευθυγραμμίστηκε με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως για παράδειγμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην πολιτική ασφάλεια, στη μακροοικονομική βοήθεια σε τρίτες χώρες, στο Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις και την υποστήριξη στην Παλαιστίνη. Τίτλος 5, διοικητικές δαπάνες. Ε, εδώ έχουμε μία μικρή μείωση κατά 31 εκατομμύρια, το οποίο δεν θα επηρεάσει την αγαστή λειτουργία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το Συμβούλιο άλλωστε δεν έχει τροποποιήσει το διοικητικό προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ε, θα επακρυπνεί όσον αφορά την επίτευξη της μείωσης ε, του ε, προσωπικού κατά 5% μέχρι το 2017 όπως προβλέπετε. Αποφασίστηκε και μία ε, συνεδρίαση στον τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό στα τέλη Ιουλίου για να συζητήσουμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία το θέμα αυτό. Ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επειδή ακριβώ συνειδητοποιούμε τι μελλοντικέ προκλήσει, κυρίω στο μεταναστευτικό τομέα και δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποιες ε, εντάσει και συγκρούσει οι οποίε ε, ε, κορυφώνονται ε, στη γείτονα περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας ισορροπημένος και υπεύθυνο ε, συμβιβασμός που μας επιτρέπει να έχουμε και κάποιο περιθώριο ελιγμών για να αντιμετωπίσουμε κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να επιδεινωθούν και αυτό είναι προφανές. ο προπολογισμό λοιπόν αποτελεί ένδειξη εσωτερικής και εξωτερικής αλληλεγγύης, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας αποσχολεί όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Κρέτσου, εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι. Καταρχήν ευχαριστήσω τον ε, Υπουργό κύριο Γραμμένια, για την παρουσίαση εκ μέρους του Συμβουλίου της, ε, των αποφάσεων του Συμβουλίου για τον 2016. Συμφωνούμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία και η υγιής διαχείριση είναι αυτό που περιμένουν οι λαοί μας. Βέβαια, οι πολίτες μας περιμένουν επίσης ε, να αντιμετωπίσουμε και επίγουσες ε, ανάγκες σε καιρούς κρίσης. Ο πρόεδρος Γιούνκερ αύριο ε, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης θα μιλήσει για το θέμα της κρίσης των προσφύγων για τι τελευταίε εξέλιξει στον αυτοκομικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χτε ε, μια δέσμη μέτρων ε, υπέρ των αγροτών. Οι οικονομικές ε, συνέπειες του μεταναστευτικού θα αντιμετωπιστούν μέσω μια τροποποιητική επιστολής τον Οκτώβριο που θα περιλαμβάνει ένα πρόσθετο πλεόνασμα στον αγροτικό τομέα εκτός των άλλων. Να σας πω τι προτείνει η Επιτροπή μας. Η Επιτροπή για το 2016 προτείνει ένα, ένα σχέδιο προπολογισμού με συγκεκριμένες πολιτικές ε, προτεραιότητες υπέρ των θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης, ε, το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, ε, για την βελτίωση των ικανοτήτων μας να απαντήσουμε στο πρόβλημα των μεταναστών και να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Η πρότασή μας αφήνει ένα περιθώριο 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποχρεώσεις και 1,6 δισεκατομμύρια σε πληρωμές και συνολικά η πρότασή μας για τον προορισμό 2016 είναι μια πρόταση ε, ενός υπεύθυνου προπολογισμού που αντιμετωπίζει πολλές ανάγκες Ευρώπης με προβλέψεις για ε, απρόβλητα γεγονότα. Ε, σέβεται τον, την συμφωνία για τις, ε, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Καλωσορίζουμε την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου για, για τα προγράμματα ε, συνοχής ε, του τίτλου 1β. Μας ανησυχούν όμως οι μειώσεις που προτείνονται σε συγκεκριμένες γραμμές του υπολογισμού σε διάφορους τομείς. Η πρότασή μας είχε ως σκοπό να μετριάσει τις ελλείψεις ε, πληρωμών των ε, περασμένων ετών και ε, για πολλές γραμμές του προπολογισμού που, που προτείνονται ο οι ανάγκες έχουν αλλάξει ασίες με πέρσι για παράδειγμα στον τομέα 4 ως αποτέλεσμα δεν, δεν υπάρχει λόγος μειώσεων σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις χαιρόμαστε που δέχεται το Συμβούλιο της Προτάσης μας για τη μετανάστευση. Σημαντικές δράσεις έχουν ήδη αναλυθεί το 2015 για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει στο μεταναστευτικό. 23 ε, πολυετή εθνικά προγράμματα ασύλου, μετανάστευσης και ολοκλήρωσης ε, έχουν εγκριθεί και 205 εκατομμύρια ε, ευρώ βοήθειας έχουν προχρηματοδοτηθεί. και 183 εκατομμύρια για το Ταμείο Συντερική Ασφάλειας. Αυτά τα χρήματα θα ρεύσουν σύντομα. Για το 2016 προτείνουμε μια συνέχιση, μέσω του, ε, συνέχιση του τροποποιητικού προπολογισμού του 2015 σε ό,τι αφορά το τίτλο 1α για την ανάπτυξη και την απασχόληση δεν συμφωνούμε με, τις, το σκεπτικό για τις μειώσεις στον ορίζοντα 2020 ε, ή το πρόγραμμα συνδέοντας στην Ευρώπη. Ε, όλα αυτά ήταν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, αποτελούν τμήμα του Ταμείου Στατικών Επενδύσεων. Το τομέας 4 βλέπει μειώσεις στα προγράμματα μας για την πολιτική γειτονία και την, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, όλα αυτά δεν θα συνεισφέρουν, αυτέ οι σημειώσει δεν θα συνεισφέρουν ε, στην σταθερότητα στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τι διοικητικέ δαπάνε, για χρόνια οι Κομισιόν και άλλα όργανα ε, έχουν αυτοπεριοριστεί και διαχείριζονται με γη τρόπο τον προπολογισμό τους. Ε, ήδη προσπαθούμε να μειώσουμε κατά 5% τα επόμενα 5 χρόνια τον προπολογισμό του προσωπικού μας. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η, αν η Κομισιόν δεχτεί τη μείωση 19 εκατομμυρίων ευρώ που προτείνει το Συμβούλιο θα έπρεπε ε, να παγώσει 206 θέσεις εργασίας συν το 4% μείωση προσωπικού που θα πρέπει να επιτευχθεί με το 2016. Ε, το προσωπικό έρευνας ε, θα επηρεαστεί σε όλα τα... και αυτό θα επηρεάσει με τη σειρά του την εφαρμογή πολλών προγραμμάτων. Τώρα για τη διαδικασία. Μέσα, μέσα Οκτωβρίου η Κομισιόν θα υποβάλει μια τροποποιητική επιστολή για την ε, γεωργία και το, νέο πακέτο, και το νέο πακέτο μεταναστευτικό πακέτο. Μέχρι το τέλος της ε, ε, περίοδο ε, συνδιαλλαγής ελπίζω θα βρούμε, ε, μια, θα βρούμε μια λύση. Ο κ. Φερνάντες. ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε, Επίτροπε, εκπρόσωποι, ε, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο είναι ε, ενωμένο ε, έχει πολύ σαφή εντολή και έχει εκδώσει πολλά ψηφίσματα. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Ε, εμείς είμαστε συνεπείς με τις προτεραιότητες μας. Στηρίζουμε την, το επιχειρηματικό πνεύμα, τις επιχειρήσεις, την απασχόληση, ε, την αλληλεγγύη εσωτερική και εξωτερική. Όλα αυτά αποτελούν τμήμα των προτεραιοτήτων μας. Και αυτό έχει συγκεκριμένε συνέπειε. Συνέπειε και στον τίτλο 1α και στο πρόγραμμα Ορίζοντα 2020, στο, στην ε, Μηχανισμό Σύνδεδας στην Ευρώπη, στην Πρωτοβουλία για την Ενική Επασχόληση κλπ. Και α μην ξεχνάμε ότι από πλευρά μα δεν δείχνουμε καμία την παραμικρή υποκρισία. Όπως σα έλεγα, όπως σας είπα προηγουμένως, είμαστε συνεπείς με τις προτεραιότητές μας. Ε, ε, λαμβάνουμε υπόψη το μεταναστευτικό, το πρόβλημα των προσφύγων και ο προϋπολογισμός μας θα πρέπει ε, να δώσει απάντηση με έργα και όχι μόνο με πράξεις σε αυτά τα προβλήματα. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε λόγια. στον τομέα 4 Έχουμε προγράμματα και μέσα που αφορούν το μεταναστευτικό και εκεί το Συμβούλιο μειώνει τον προϋπολογισμό κατά 350 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές. Στον τομέα 4 έχουμε το, προ, το προενταξιακό μηχανισμό και εκεί έχουμε μείωση. Ε, η, ε, μειώνεται κατά πάνω από 100 εκατομμύρια, ευρώ ε, ο προϋπολογισμός του, ε, της πολιτικής γειτονίας ο μηχανισμός για τη συνεργασία για την ανάπτυξη ε, μειώνεται κατά 143 εκατομμύρια ευρώ. Επίση το Συμβούλιο περικόπτει συνολικά 1,4 ε, δισεκατομμύρια ευρώ από την πρόταση τη Κομισιόν. Το Συμβούλιο <laughs> ενδεχομένω έκανε σύγκριση με τον προπολογισμό του 1980 και του 1990, όχι με τον προπολογισμό του 2015. Μας λέει ότι εγκρίθηκε ομόφωνα ε, το, το ε, χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τα προηγούμενα έτη. Όμως το Συμβούλιο είχε ήδη μειώσει τον προπολογισμό και τώρα κάνει περισσότερες ακόμα μειώσεις και περικοπές. Αυτό είναι ακατανόητο, ασυνεπές, έρχεται σε αντίθεση με τις ίδιες τις προτεραιότητες και τις προτάσεις του Συμβουλίου στο παρελθόν. Το Συμβουλίο δεν μπορεί να μας λέει, και τελειώνω, τέσσερα λεπτά όμως μου είχαν δοθεί οι Πρόεδρε, το Συμβουλίο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μειώνει μόνο τις γραμμές που υπάρχει υψηλή ε, απορροφητικότητα. Ε, γιατί περικόπτει το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη, περικόπτει το ορίζοντας 2020 περικόπτει μέσα τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι να τον ισχύεται τέτοια πράγματα το Συμβούλιο. Εδώ, στην αίθουσα της Ολομέλειας. Λίγο ντροπή πρέπει να νιώσει το Συμβούλιο. Γιατί όλες αυτές οι δηλώσεις, όλα αυτά τα λόγια δεν έχουν καμία σχέση με παλιότερε δηλώσει και αποφάσει του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Φερνάνδη. Τρία λεπτά είχατε. Τόσο λεπτό χρόνο όσο και ο κύριο Ντεπρέ, τον οποίο δίνω τώρα το λόγο. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τέσσερα είπατε έτσι. Ναι, με συγχωρείτε για το αστείο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, συμμερίζομαι την ανακούφιση που εκφράζεται για το 2015 και το 2016 ιδιαίτερως όσον αφορά τις πιστώσεις των πληρωμών. Πέρυσι είχαμε περίπου περάσει τις διαπραγματεύσεις της Δημοσιονομικής Αρχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό του ουσιαστικά για να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα των πληρωμών. Τώρα δεν είναι καλή η κατάσταση το 2015. Είναι κακή αλλά σταθεροποιείται και θα βελτιωθεί για το 2016. Δεν θα κρατήσει όμως αυτό γιατί μέχρι το τέλος των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών θα χρειαστεί να ανέβουν και μάλιστα ριζικά οι πιστώσεις των πληρωμών. Γιατί, γιατί διαρθρωτικά δεν έχει γίνει τίποτα για να βελτιωθεί η κατάσταση ενώπιον της οποίας θα βρεθούμε πριν το τέλος των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών. Για τον προπολογισμό 2016, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε τρεις μεγάλες προτεραιότητες την ανάγκη να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, να συνδυάσουμε ανθρωπισμό και αποτελεσματικότητα όσον αφορά τους πρόσφυγες που αναζητούν ασφάλεια και άσυλο στις χώρες μας. Και τρίτη μεγάλη προτεραιότητα που λησμονήσατε σήμερα, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν ηθελημένο, την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την δημοκρατική απειλή που ε, ρίχνει βαρύ τον ίσκιο της. Δεν θα αναφερθώ στην τρίτη αυτή πρόκληση παρά μόνο για να υπενθυμίσω ότι πρέπει να ενισχυθεί το ανθρώπινο και υλικό δυναμικό να διατεθούν στα κοινοτικά όργανα όπως η Europol, η Eurojust, η EULISA ε, που διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών, τα μέσα για την καταπολέμηση της δημοκρατίας και την αποτροπή επανάληψης τρομοκρατικών επιθέσεων. Θεωρούμε ότι τα μέσα τα οποία έχετε προβλέψει σε επίπεδο Συμβουλίου αλλά και σε επίπεδο Επιτροπής πρέπει να πω δεν αρκούν για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητα αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των οργάνων και υπηρεσιών. Όμως ε, η μεγαλύτερη πρόκληση και ο κίνδυνος και το διακύβευμα είναι αυτό της ε, προσέλευσης ε, της μαζικής εισρωής προσφύγων προς την Ευρώπη, το είπε και ο πρόεδρος Κλώτης Γιουνκέρ, ε, έναντι των πολιτικών ε, υπευθύνων των κρατών μελών με τους οποίους συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και δεν αναφέρομαι εδώ στον κύριο Ορμπάν. Αλλά θα ήθελα να πω τα εξής κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου ότι για το 2016 όντως αναφέρεται μια αύξηση 169 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2015. Αλλά δεν αρκούν αυτά και δεν θα αρκέσουν ποσού δε μάλλον καθώς το κόστος για την κατανομή των προσφύγων θα σημαίνει σημαντικές αυξήσεις. Εάν θέλει 120.000 εθελοντέ, ο κύριος Ζων Κλοντ με τους ε, ήδη υφιστάμενους 40.000 θα χρειαστούν πάντα από 960 ε, εκατομμύρια ευρώ για να τηρηθούν οι προϋποθέσεις. Δεν έχει κλείσει λοιπόν εδώ το πρόβλημα. Μια λέξη ακόμα πρόεδρε για να ολοκληρώσω. Λυπούμε όπως και ο φίλος Χωσέ Φερνάντες που γεγονός, για το γεγονός ότι το Συμβούλιο θεωρεί πως χρειάζεται ακόμη να προσαρμόσει κάποιες δημοσιονομικές ε, γραμμές για το Connecting Europe, την ε, διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη δηλαδή και άλλες ε, τέτοιες ε, θέσεις του προπολογισμού που όμως έχουν τεράστια σημασία όπως ορίζουν 2020, 2014, 2015 για τους, οποίους, για, για τους όμως και τις θέσεις δημιουργείται τις ε, συνθήκες που δεν μπορούν να δώσουν κανένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ και για να τελειώσει αυτή η γενική συζήτηση ο κύριος Γραμμένια που ασφαλώς θα έχει να δώσει απαντήσεις. Γραμμένια. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι, η στιγμή, ότι είναι η στιγμή σήμερα να πούμε στη συζήτηση επί της ουσίας για την πρόταση του Συμβουλίου και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τους δύο εισηγητές, τους κυρίους Φερνάντες και Ντεπρέ, τους οποίους ευχαριστώ πάντως για την προσήλωση και το δυναμισμό για τον οποίο υπερασπίζονται τις διάφορες πιστώσεις. Θέλω απλώς να υπογραμμίσω πως σημειώσεις που επέφερε το Συμβούλιο γίνονται κατόπιν προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προτείνει σημαντικές αυξήσεις στα σημεία τα οποία σας ανέφερα. Στο κεφάλαιο 4, σας υπενθυμίζω, έχουμε αυξήσει τις πιστώσεις των πληρωμών της τάξης των 42 και της 100. Όταν, μιλούμε για περικο... Όταν γίνεται λόγος λοιπόν για περικοπές, οι περικοπές δεν αφορούν τον προϋπολογισμό του 2015, αλλά ε, μείωση των προταθέντων από την Επιτροπή ιδιαίτερα αυξημένων ποσών. Όπως είπα, δεν θα πούμε τώρα στη λεπτομέρεια της διαπραγμάτευσης. Χαίρομαι που άκουσα ότι παρατσύρθηκα σε λυρισμούς. Εγώ νόμιζα ότι μιλούσα σταράτα και απλά. Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά που θα είμαι μεταξύ σας να μιλήσω πιο προσγειωμένα. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι θέλουμε να δουλέψουμε με σας χέρι-χέρι. Θα ακούσουμε κάθε πρότασή σας και εγώ τίνω χείρα συνεργασίας Είναι μια συνεργασία ειλικρινή και επικοδομητική ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, συμβασμό που καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα υπάρξουν έκτακτες δαπάνες με, και λόγω των επιδεινούμενων συνθήκων θα χρειαστεί να βρεθεί, θα είναι δύσκολος συμβασμός. Ο πρόεδρος Γιουνκέρ είπε ότι η επίλυση των προβλημάτων των μεταναστευτικών δεν μπορεί να γίνει με μηδενικό κόστος. Ούτε στη γεωργία μπορούν να λυθούν τα προβλήματα, όπως είπε και η Επίτροπος. Ε, μπορούν να λυθούν τα προβλήματα εύκολα. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να κλείσει ο προπολογισμό. Η μόνη διαβεβαίωση που μπορώ εγώ από πλευρά μου να σα δώσω σήμερα είναι ότι θα παίξουμε με ανοιχτά χαρτιά και ότι θα αναζητήσουμε υπεύθυνου και ε, εφικτούς συμβιβασμούς για να κάνουμε καλή δουλειά προς τα έξω όσο και προς τα μέσα στο χώρο της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνει τη συζήτηση και πάμε στο επόμενο θέμα. Je vous propose que nous dans un tout petit, un petit instant. Très bien. Μια μικρή διακοπή, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή αλλαγή, ώστε να, έρθει ο κύριος Αβραμόπουλος.